δημόσια συνεδρία μεταδίδεται μέσω του διαδικτύου. Έχουμε ψηφοφορίες, ελπίζω να έχετε φέρει μαζί τις κάρτες. Αλλά ίσως πρώτα να κάνουμε ένα τεστ, μια δοκιμή. Περιμένω να ετοιμαστείτε. Και το μεταξύ σας επισημαίνω ότι στις 14 Νοεμβρίου, ημέρα 5η, Έχουμε την διακοινοβουλευτική συνάντηση με εκπροσώπους των αντίστοιχων υπηρεσιών των κρατών μελών για μια καλύτερη επαλήθευση των δαπανών των δημοσίων δαπανών για τις 14 Νοεμβρίου από τα Εθνικά Κοινοβούλια λοιπόν, αν έχετε συναδέλφους στους οποίους επικοινωνείτε, μπορείτε να τους επισημάνετε συνεδρία συνεδρίαση αυτή. Και βεβαίως περιμένουμε μέχρι τις 7 Νοεμβρίου για να κλείσουμε τον κατάλογο των συμμετεχόντων. Και πάω στο σημείο 3 της ημερησίας διάταξης, έγκριση πρακτικών 16-17 Σεπτεμβρίου. 25-26 Σεπτεμβρίου, 2 Οκτωβρίου. Υπάρχουν ε, παρατηρήσεις για τα πρακτικά αυτά. Όχι. Και ως εκ τούτου εγκρίνονται τα πρακτικά. Και πάμε στο σημείο 4 της μερισίας διατάξεως. Που έχει αναβληθεί. Πάμε στο σημείο 5. Εδώ ψηφίζουμε. Και παρακαλώ τον εισηγητή εάν θέλει το λόγο πριν ή μετά τη συνεδρία την προτιμάτε, μετά μάλιστα. Όχι πριν. Ευχαριστώ. Λέω ο Είναι πολύ σημαντική αυτή η έκθεση αφορά και την Επιτροπή Μεταφορών, μια που έχει σχέση με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων. Πρόκειται για την μοναδική ρυθμιστική αρχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τους σιδηροδρόμους. Θέλουμε να εγκριθούν τελικά κάποια ε, κοινά τεχνικά πρότυπα. Βεβαίως και θέλουμε να γίνεται υγιής οικονομική διαχείριση, υγιής διοίκηση αυτού του οργανισμού. Οπότε και από πλευράς Επιτροπής Μεταφορών ε, ενδιαφερόμαστε πάρα πολύ να γίνει η ψηφοφορία. Σας ευχαριστώ πολύ και έτσι περνάμε στην ψηφοφορία. Θα ήθελα να κάνουμε μια δοκιμαστική πρώτα, να κάνουμε μια επαλήθευση με τις ηλεκτρονικές μας κάρτες. Αρχίζουμε τη δοκιμή. Ψήφισαν όλοι. Δουλεύουν τα μηχανήματα. Λείπει μια κάρτα από ό,τι φαίνεται. Τώρα κλείνουμε την ψηφοφορία αυτή. 11 είναι οι παρόντες. Πέντε τέσσερις, δύο. Και έτσι μπορούμε να ξεκινήσουμε τη συνέδριαση, την ε, ψηφοφορία. Τροπολογία υπερθμών 3, υπέρ παρακαλώ, κατά άποχες. Ηλεκτρονική επαλήθευση, δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν οι πάντες. πέρασε της ψηφοφορίας.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 Έχει απορριφθεί. Τροπολογία 10 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 11 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 12 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 13 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 16 υπέρ κατά αποχές επαληθεύουμε δεν ήταν σαφές το αποτέλεσμα στη 16 άρχεται η ψηφοφορία ψήφισαν οι πάντες πέρασε της ψηφοφορίας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 αποχές εγκρίνεται 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 51 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 52 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 53 υπέρ κατά Ας επαληθεύσουμε την 53. Πέρας. Εγκρίνεται 54 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 55. Να, η 50 είχε απορριφθεί, 55 λοιπόν, υπέρ. Κατά αποχέ συγκρίνεται 56. Αποχές απερίφθη. 57 υπέρ. Κατά αποχές απερίφθη. 58 υπέρ. Κατά αποχές απερίφθη, αλλά σε παληθεύσουμε παρακαλώ. 58. Πέρασε. Εγκρίνεται. Α, όχι. Ε, απερίφθη. Λόγω ψηφία. 59 υπέρ. Κατά αποχές απερίφθη. Ποια έχει αποσυρθεί. Όχι, είναι αργότερα. 31 υπέρ. Κατά αποχές συγκρίνεται. 60 υπέρ. Κατά αποχές απερίφθη 61 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 62 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 63 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 22 υπέρ κατά αποχές δεν σε το αποτέλεσμα σε την 22 παρακαλώ 23 τώρα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 64 υπέρ, α, έχει αποσυρθεί. 65 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 66 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 24 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 25 υπέρ, κατά αποχές απερίφθη. 26 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 27 υπέρ, κατά αποχές απερίφθη, 28 υπέρ, κατά αποχές. Ας επαληθεύσουμε την 28. Πέρασε φορέας. Μπάρ τη υπέρ κατά αποχή. Καλά. Επομένω εγκρίνεται. 29 υπέρ κατά άποχες. Ας επαληθεύσουμε, γιατί πιστεύω ότι έχει απορριφθεί, αλλά 29 ε, λοιπόν, επαληθεύση. Πέρας. Κύριε Γκρέσλε, ο κύριος Χόισλινγκ, εγκρίνεται επομένως. Υπαριθμόν 1 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 30 υπέρ. Κατά. Αποχές το επαληθεύουμε. 32 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 33 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 34 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 35 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη προτείνεται να ψηφίσουμε από την 36 ως τη 42. Συμφωνείτε όλοι. Ομού. 36 ως 42. Ομού. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απερίφθησαν. Τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 43 υπέρ κατά αποχές απερίφθη, 44 υπέρ κατά αποχές απερίφθη ή 45 πίπτη. Στο σύνορο τώρα ηλεκτρονική ψηφοφορία παρακαλώ. Πέρας. Για να σε ότι Τρεις επιπλέον υπέρ. Σημειώνουμε. Ευχαριστώ πολύ και συγχαρητήρια στον κύριο Λιμπεράτης και τον εισηγητή. Και έτσι τώρα Ja, meine Damen und Herren, ich komme zum nächsten. Και έτσι περνάω στο επόμενο θέμα Θεωρήσαμε να περιλάβουμε το θέμα αυτό στην ημερήσια διάταξη. Καλωσορίζω τον κύριο Νίβεν Μάτε μέρο του Λεκτικού Συνεδρίου. Εδώ είστε. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν θερμά. Και παρακαλώ πρώτα την εισηγήτρια να μας πει αν θέλει να λάβει το λόγο. Παρακαλώ. Θα θέλατε να κάνετε κάποιες εισαγωγικές παρατηρήσεις. Καλώς. Τότε θα επισημάνω, κύριε Μάρτες, ότι σας ε, παρακαλέσαμε να λάβετε για μια φορά το λόγο εδώ ενώπιον της Επιτροπής. Ναι, πολύ καλό να έρθετε εδώ μπροστά. Σας ευχαριστώ. Σα Σας καλέσαμε λοιπόν για άλλη μια φορά στην Επιτροπή μας κύριε Μάτες. Γιατί θέλαμε να συνομιλήσουμε και πάλι μαζί σας. Σας ε, ακούσαμε σε μια πολύ εντατική ακρόαση κατά την παρουσίαση των υποψηφιωτήτων ε, ως υποψήφιο μέλος του Λαγκτικού Συνεδρίου μας είχατε καταθέσει και μια επιστολή όπου δεσμευόσασταν πως σε περίπτωση ε, αρνητικής ψηφοφορίας πλευράς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν θα αναλαμβάνατε καθήκοντα. Αυτή ήταν και η αρνητική ψήφος την οποία έδωσε η Ολομέλεια του Κοινοβουλίου. Και διαρωτώμεθα πώς ε, εξηγείται η απόκληση μεταξύ των δηλώσεών σας εδώ, σε αυτό το όργανο, την Επιτροπή μας, που έγιναν μάλιστα και γραπτός, οι διαβεβαιώσεις που δόθηκαν γραπτός, ότι δεν πρόκειται να αναλάβετε καθήκοντα, και βέβαια η ε, στάση που εν τέλει τηρήσατε. Ξέρετε ότι αυτό, φαντάζεστε ότι αυτό δεν είναι κάτι το οποίο εμείς ως Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού παίρνουμε, ε, αντιμετωπίζουμε με ελαφρότητα. Παρακαλώ να λάβετε το λόγο λοιπόν. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας στην ε, νέα αυτή ακρόση που μου δίνει τη δυνατότητα να εξηγήσω δημοσίως και προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για ποιο λόγο δεν απέσυρα την υποψηφιότητά μου από το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο. Θα ξεκινήσω ευθύ αμέσω λοιπόν για ποιο λόγο έπραξα τα όσα έπραξα. Μετά την πρώτη ακρόαση του Μαΐου έλαβα ένα επίσημο ερωτηματολόγιο το ερωτηματολόγιο το οποίο αποστέλλεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προς όλες τους υποψήφιους για το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο. Η τελευταία ερώτηση είχε να κάνει με το πώ θα αντιδρούσα σε περίπτωση αρνητική γνωμοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ω προ αυτό είπα ότι ήταν αρκετά πιθανό να αποσύρω την υποψηφιότητά μου, εξετάζοντα πάρα πολύ προσεκτικά του λόγου που έχουν οδηγήσει στην αρνητική αυτή γνωμοδότηση. Ωστόσο δεν είχα λάβει και δεν θα λάμβανα μια τελική απόφαση για το ζήτημα αυτό, αν δεν άκουγα πρώτα τις αντιρρήσεις που υπάρχουν και που εκφράζονται για, τη δική μου την, για το δικό μου το διορισμό. Σας είπα ότι ενδεχομένως κατά πάσα πιθανότητα να απέσυρα την υποψηφιότητά μου. Θεωρούσα ότι αν δεν ήμουν σε θέση να απαντήσω σε κάποιες από τις ερωτήσεις για τα επαγγελματικά μου προσόντα, τις οποίες θέστε κατά τη διάρκεια της ακρόασης, όντως θα απέσυρα την υποψηφιότητά μου. Η ακρόαση αυτή έλαβε λοιπόν χώρα και μετά την ακρόαση αυτή ανέλησα πάρα πολύ προσεκτικά όλες τις παρατηρήσεις που γίνανε από τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου του Προπολογισμού και πραγματικά εκτιμώ ιδιαίτερα κάποια θετικά σχόλια τα οποία ακούστηκαν για τα επαγγελματικά μου προσόντα. Ήδη χθε τα ξαναδιάβαζα και θεωρώ ήταν ιδιαίτερα θετικά. Κατέγραψα όμως και τις παρατηρήσεις εκείνες που είχαν να κάνουν με την απώλεια άμεσης ή μάλλον την απουσία άμεσης εμπειρίας όσον αφορά τον δημοσιονομικό έλεγχο. Επίσης, κατά τη διάρκεια των επόμενων εβδομάδων ακούστηκαν κάποιες ε, παρατηρήσεις, σύμφωνα με τις οποίες κατέληξε το συμπέρασμα ότι ε, η Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού είχε καταψηφίσει τη δική μου την υποψηφιότητα, χωρίς όμως να φαίνεται τελικά ότι υπήρχαν κάποια προβλήματα αξιοκρατικά, ότι θα έπρεπε δηλαδή για λόγους αξιοκρατικούς να αποσύρω την, την υποψηφιότητά μου. Πρέπει να σας πω ότι ε, μου κάνει εντύπωση το ότι συμπεριλάβατε στο επίσημο ερωτηματολόγιο την ερώτηση αυτή που είχε να κάνει με το πώς θα αντιδρούσα σε περίπτωση αρνητικής γνωμοδότησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θεωρώ ότι είναι κάπως περίεργο να έπρεπε εγώ εμέσως να δεσμευτώ ότι θα τηρήσω την ε, γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προκειμένου να κερδίσω και τη δική σας την ε, εύνοια. Ξέρετε επίση ότι ε, σύμφωνα με τη συνθήκη λειτουργία Ευρωπαϊκή Ένωση, το Συμβούλιο είναι αυτό το οποίο παίρνει τελική απόφαση. Στην γραπτή μου λοιπόν απάντηση αναφέρομαι στου υφιστάμενου κανόνε για το διορισμό στο λεκτικό συνέδριο, κανόνε που απορρέουν από την ίδια τη συνθήκη. Κατά τη διάρκεια τη ακρόαση όμω υπήρχαν πάρα πολλοί που επέμεναν να απαντήσω αυτή την ερώτηση. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ περίεργο ότι τελικά η ερώτηση αυτή έγινε η πιο σημαντική ερώτηση κατά τη διάρκεια τη ε, ακρόαση. Θεωρώ πάντως ότι σας έδωσα αρκετές πληροφορίες στα πλαίσια της γραπτής μου απάντασης και είπα πάρα πολλές φορές ότι εγώ δεν μπορώ να αλλάξω, να τροποποιήσω τους κανόνες που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το διορισμό των μελών του ελεκτικού συνεδρίου. Είναι κανόνες οι οποίοι παγιώνονται στα πλαίσια της συνθήκης. Απαντώντας λοιπόν κάποια στιγμή στην ερώτησή σας, αφού επιμείνατε πάρα πολύ, είπα ότι σε περίπτωση που καταψηφίσετε τελικά την γνωμοδότησή την υποψηφιότητά μου, συγχωρείτε, και αφού επιμένετε τόσο πολύ, ενδεχομένως να αποσύρω την υποψηφιότητά μου. Θεωρώ πάντως ότι η δέσμευση αυτή την οποία άτυπα έδωσα στο Κοινοβούλιο την επανέλαβα και σε μια επιστολή της 5ης Ιουνίου. Είπα όμως τότε, στην επιστολή αυτή, ότι Κατά τη διάρκεια της ακρόασης είπα πάρα πολλές φορές ότι δεν μπορώ εγώ να τροποποιήσω τους κανόνες και ότι ήθελα να δώσω εμέσως ένα μήνυμα προς την Επιτροπή ελέγχου του προπολογισμού, η οποία φαινόταν ότι ήθελε να τροποποιήσει τους κανόνες διορισμού στο ελεκτικό συνέδριο. Και είχα πει ότι δεν θα μπορούσε σε καμία περίπτωση μια τέτοια τροποποίηση να αποτελέσει προϋπόθεση για την υποστήριξη ενός υποψηφίου. Ένας υποψήφιος θα πρέπει να κρίνεται βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων και όχι βάσει της προϋπόθεσης αυτής. Στη συνέχεια το Κοινοβούλιο καταψήφισε την ε, υποψηφιότητά μου. Ανέλησα την απόφασή σας αυτή και κατέληξα στην απόφαση ότι ε, είχατε επιμείνει πάρα πολύ στην έμεση αυτή δεσμευσή μου για να αποσύρω την υποψηφιότητά μου και ότι ε, η αιμονή σας αυτή τελικά δεν είχε να κάνει τόσο με τα αξιοκρατικά κριτήρια διορισμού όσο με το ότι θέλατε εγώ να συμμορφωθώ πάση θυσία στην ε, αρχική μου δέσμευση. Τελικά όμως το Συμβούλιο με διόρισε σαφώς τα πράγματα θα μπορούσαν να είχαν εξελιχθεί διαφορετικά. Θα ήταν πολύ καλύτερο να μην είχα κάνει τη δήλωση αυτή κατά τη διάρκεια της ακροασής σας και να είχα μείνει στην αρχική μου τοποθέτηση. Ζητώ συγγνώμη αν προκάλεσα σύγχυση σε κάποιους. Σε καμία περίπτωση δεν ήταν πρόθεσή μου να παραπλανήσω κανέναν, είτε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε αλλού. Ω μέλο λοιπόν του Ελεκτικού Συνεδρίου θέλω να συνεχίσω να καταβάλω τι προσπάθειε τι οποίε καταβάλω για να έχουμε μια επικοδομητική συνεργασία με την Επιτροπή σα για να πετύχουμε κάποιου κοινού στόχου. Ελπίζω ότι δεν θα βασιστούμε αυτή τη στιγμή σε κάποιες παρανοήσεις στη μελλοντική μας συνεργασία. Ελπίζω να αλλάξετε προσέγγιση και να μπορέσουμε να συνεργαστούμε από κοινού προκειμένου να εξυπηρετήσουμε όσο δυνατόν πιο επικοδομητικά τα συμφέροντα των Ευρωπαίων πολιτών όσον αφορά την καλύτερη δυνατή διαχείριση των κοινοτικών πόρων. Για άλλη μια φορά επαναλαμβάνω ότι θέλω να δημιουργήσω συνθήκες επικοδομητικής συνεργασίας με εσά. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Μάρτες. Τώρα παρακαλώ την εισηγήτρια μου, αν θέλει να λάβει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Μάτες που ήρθατε να μας ε, μιλήσετε, να αυτοσυστηθείτε ούτως υπήν για δεύτερη φορά στην Επιτροπή μας. Και θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι όντως μας συνεκλώνησε, μας εξέπληξε η απάντηση γιατί γνωρίζετε ότι για την Ευρωπαϊκή Οικοδόμηση το Κοινοβούλιο και κάθε θεσμικό όργανο ε, βάζει το λιθαράκι του όσον αφορά την ισορροπία των δυνάμεων, την εκπροσώπησή του και εμείς από τις θέσεις μας ως δημοκρατικά εκλεγμένο σώμα πρέπει να συνεργαστούμε με το ελληνικό συνέδριο και πρέπει επομένως να δούμε τους, ε, ε, τους, τους υποψηφίους και εν πάση θα πρέπει να είναι ουσιαστική αυτή η ερωταπάντηση που γίνεται για να είμαστε σε κάποιο είδους σχέση εμπιστοσύνη με αυτούς τους συμβούλους του ελεγκτικού συνεδρίου. Και σε πολλές περιπτώσεις είμαστε συνομοθέτες. Οπότε η Επιτροπή μας του Δημοσιονομικού Ελέγχου αυτή τη στιγμή είναι στην πιο κατάλληλη θέση, ε, αναλαμβάνοντας τις ευθύνες της, έναντι του Συμβουλίου και έτσι τα πράγματα έχουν περιπλακεί αρκετά. και κατά κάποιο τρόπο έχουμε έρθει σε αντιπαράθεση τώρα με το Συμβούλιο. Να σας πω όπως λοιπόν τα πράγματα ως ε, βουλευτήνα ότι κάπως υπερβολικά μπορώ να πω ότι εμείς χρησιμοποιούμε αυτή την ερώτηση και όπως λέτε και εσείς κρυπτό να γίνει η απόφαση και η ψηφοφορία, αλλά αυτό, αυτό εν μέρει έχει σχέση με το ότι εμεί είμαι θέση θέση να αλλάξουμε, να ανατρέψουμε της υποψηφιότητας ε, που κατεβάζει το Συμβούλιο για το Ελληνικό Συνέδριο. Πολλές φορές όμως είναι αλήθεια ότι οι υποψηφιότητες που κατεβάζει το Συμβούλιο δεν έχουν καμία σχέση με αυτό το οποίο ζητεί, απαιτεί το κοινοβούλιο αυτό ως υποψηφιότητες. Επομένως με αυτόν τον τρόπο λέμε ότι έχουμε το κλειδί ούτως ώστε να εξασφαλίσουμε το ότι ο υποψήφιος οποίος κατεβαίνει παρουσιάζεται εδώ ε, ως ε, υποψήφιο μέλος του Ελληνικού Συνεδρίου μπορεί να αποσπάσει την απόλυτη ε, εμπιστοσύνη του Κοινοβουλίου της Πλειοψηφίας αυτού. Μα γι' αυτό σας λέω ότι πρόκειται για πολύ σημαντική διαδικασία οπότε να τι ισχύει ως προς εμάς και το Συμβούλιο άλλη σχέση δική σας με το Συμβούλιο άλλη με την Επιτροπή μας και το Κοινοβούλιο. Οπότε γι' αυτό σας είπα ότι στην επιστολή σας μας προκάλεσε ε, μεγάλη έκπληξη ε, ε, αυτά που λέτε ως συστάσεις και ότι τι θα γίνει αν το Συμβούλιο δεν υποστήριξει την υποψηφιότητά σας. Άλλωστε τα είπαμε και τα ξαναείπαμε κατά την πρώτη ακρόαση. Και αυτά που λέτε εσείς για την ενδεχόμενή σας παρέτηση. Είπατε ότι υποβάλλετε την παρατησία σα στην κυβέρνησή σα δεν έγινε αποδεκτή. Εντάξει, τι να σα πω. Ε, σας πιστεύουμε όπω και εσεί μα πιστεύετε. Τι να, δεν ξέρουμε τι λεπτομέρειε και τι έγινε. εσεί τα ξέρετε. Εσείς ούτως ή άλλως πρέπει να τηρήσετε ε, το λόγο σας σε σχέση με αυτήν την διατύπωση του ενδεχομένου της παρέτησης. δεν σας φάνηκε φυσιολογικό το ότι εμείς έχουμε αυτή την αντίδραση σε σχέση με αυτό το εκ των υστέρων σύστημα σύμφωνα με το οποίο ζητείται αιτιολόγηση της δικής μας απόφασης. Έχει γίνει μια σειρά ενεργειών για αυτή τη διαδικασία. Δεν λέμε ότι όλοι συμφωνούμε με όλες. Αλλά, όπως είπαν και οι συνάδελφοι, είναι ενδιαφέρον το, το ότι θα πρέπει οι υποψήφοι να καταλάβουν τι γίνεται σε σχέση με την απόφαση που εμείς λαμβάνουμε. Να μας ρωτήσουν για αυτή την απόφαση. Κανένα πρόβλημα να την επεξηγήσουμε και αιτιολογήσουμε. Όμως κατανοείτε ότι τώρα δυσκολευόμαστε έτσι όπως το έχετε θέσει μας λέτε για μια παρέτηση, δεν ξέραμε τίποτα, λέτε δεν έγινε αποδεκτή και λέτε ότι όλα αυτά ισχύουν έως ότου εμείς επιβεβαιώσουμε την επιλογή και εκλογή σας. Σας ακούσαμε, σας ακούσαμε. Εσείς τηρείτε το λόγο σας. Όλα αυτά είναι θεμητά. Δεν σας κατηγορούμε. Άλλωστε και με τη δουλειά μας κάνουμε που βάλουμε τις ερωτήσεις που χρειάζεται το κοινοβούλιο για να μπορέσει να λάβει μια απόφαση. Οπότε, εσείς τώρα με τη σειρά σας έχετε κάτι να πώς αγάγετε ούτως ώστε να μας πείσετε σε σχέση με το διορισμό σας, την παρέτηση, σε σχέση με όλα αυτά. Για να μας πείσετε dazu antworten, Herr bitte. Παρακαλώ, κύριε Μάθες, για να απαντήσετε. Ναι, κύριε Πρόεδρε. Θα σα το πω ως Έγραψα την επιστολή μου, απόσυρση υποψηφιότητα, την υπέγραψα και πήγα να συναντήσω τον Πρωθυπουργό, ο οποίο μου ζήτησε να μην αποσυρθώ από τη διαδικασία. Και έτσι απεφάσισα να παραμείνω στη διαδικασία. Και απέστειλα επιστολή στον πρόεδρο του Κοινοβουλίου, την οποία όμως δεν έστειλα διότι δεν έχει θέση στη διαδικασία, δεν προβλέπεται. Τώρα, εάν μου επιτρέπετε, θα πρότεινα να αφήσουμε κατά μέρος τις παρεξηγήσεις αυτές. Στο έργο μου, ε, ως μέλος της, ε, του ελεγκτικού συνεδρίου θα έρχομαι συχνά να σας επισκεφθώ, να συνομιλήσουμε και θα κάνω ό,τι μπορώ για να επιδείξω πνεύμα συνεργασίας και τις βέλτιστες δυνατές σχέσεις μαζί σας. Και θα κάνω ό,τι μπορώ για να σας πείσω ότι ήμουν καλός υποψήφιος και όταν καλή η επιλογή του προσώπου μου για την θέση αυτή. Αυτό θα προσπαθήσω να το κάνω στη συνεργασία μαζί σας. Ο κύριος Μιούλτερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Νομίζω ότι μετά τη δήλωση αυτή γίνεται χειρότερη η κατάσταση. Τι να πιστέψουμε. Εσείς δηλαδή μας λέτε ότι η ψηφοφορία στην οποία ε, προέβημε δεν είχε να κάνει με τις δεξιότητες σας αλλά με το κατά πόσον θα δεσμευόσασταν να αποσύρετε την υποψηφιότητά σας μετά την ψηφοφορία. Πού το ξέρετε εσείς, δηλαδή μπορείτε να διαβάσετε τι σκέπτονταν οι 396 που σας καταψήφισαν. Εγώ σας διαβεβαιώ ότι δεν ήταν καθόλου σημαντική αυτή η δέσμευση στην ψηφοφορία και αφορούσε κυρίως τις ε, ικανότητές σας, τα προσόντα σας τα οποία κρίθησαν ανεπαρκή. Την ερώτηση αυτή την έχουμε κάνει και σε άλλους υποψηφίους, την κάνουμε παγίως και υπήρξαν και άλλοι υποψήφοι στο παρελθόν, οι οποίοι είχαν πει ότι θα αποσυρθούν αν ε, λάβουν αρνητική ψήφο και τελικά τήρησαν την υπόσχεση αυτή τη δέσμευση. Εσύ είσαι το μόνος ο οποίος δεν τήρησε τη δέσμευσή του. Δεν ξέρω τι είδου ε, σχέση μπορούμε να έχουμε στην Κροατία εάν ε, οι αξιωματούχοι μπορούν να ε, παραβιάζουν δεσμεύσεις που έχουν λάβει ενώπιον του Κοινοβουλίου με τέτοια ευκολία. Πάντως, εγώ, από αυτά που βλέπω, είστε κακός, θα είσαστε κακός μέλος για το ελεκτικό συνέδριο και κακός εκπρόσωπος της Κροατίας. Έχουμε σοβαρές επιφυλάξεις για τις ε, ικανότητές σας και επιπλέον δεν είπατε την αλήθεια στο κοινοβούλιο. Και αυτό για μένα δεν σας καθιστά άξιο μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου. Κατάσταση είναι ότι κανείς δεν μπορεί να σας απαλλάξει των καθηκόντων σας, μόνο εσείς μπορείτε να το πράξετε αυτό, αλλά δεν πρόκειται κανείς από το κοινοβούλιο στα επόμενα χρόνια να σας πιστέψει σε οποιαδήποτε έκθεση εκδώσετε και υπογράψετε. Κύριε Μίλτερ, ευχαριστώ. Θέλετε να δώσετε απάντηση αμέσω ή περιμένετε να ακούσετε άλλη μια ερώτηση πρώτα. Κύριο Σοντή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι ατυχής αυτή η υπόθεση και θα ήθελα να την κλείνουμε. Γιατί μας λέτε κύριε Μάτες ότι δεν αλλάζετε εσείς τους κανόνες της συνθήκης και έχετε δίκιο σε αυτό. Ε, λέτε ότι δεν μπορεί η Επιτροπή του Ελέγχου του Προπολογισμού να τροποποιήσει τους κανόνες. Έχετε άδικο σε αυτό. Τους κανόνες μπορούμε να τους αλλάξουμε εμείς γιατί πρόκειται για δικαίωμα πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μπορεί να ζητήσει αλλαγή των ε, συνθήκων. Και τέλει, κύριε Ρεμάτες, ε, μας βολεύει αυτό που κάνατε. Γιατί εμείς δεν ε, την έχουμε στημένη σε κανέναν εν γέννη. Ε, ε, με εσά τα έχουμε, διότι δεν τηρήσατε τη δέσμευση για απόσταση τη υποψηφιότητά σα. Και από ό,τι μα λέτε, αυτό έγινε για τη συστολή του Πρωθυπουργού σα. Δηλαδή δεν ήσταν εξάρτητο απέναντι στην κυβέρνησή σα. Εκεί που λέτε δηλαδή στην κυβέρνηση ότι θέλετε να αποσύρετε την υποψηφιότητα, ο Πρωθυπουργό σα λέει όχι, όχι, θα μείνει και εσεί υπακούετε σε αυτέ τι εντολέ του Πρωθυπουργού. Άρα λοιπόν, ε, πραγματικά τα έχουμε μαζί σας, αλλά θα γυρίσουμε σελίδα που ζητάτε. Αλλά τι τα έχουμε πραγματικά με την κυβέρνησή σας, με τον πρωθυπουργό σας, ο οποίος όφιλε να έχει κοιτάξει τις απόψεις που, εκφρα... εξέφρασε το Κοινοβούλιο και να μην ζητούσε από το Συμβούλιο να επικυρώσει την ε, υποψηφιότητας, ε, ξέρουμε πολύ καλά τι κάνουν ε, τα μέλη του Συμβουλίου με τους πρεσβευτές τους. Είναι με το Δουνέ και Λαβίν όλοι. Από την ώρα που λέει ο Πρωθυπουργός ο δικός σας, θέλω τον κύριο Ματές γιατί ο ελεγκτικό συνέδριο, βεβαίως ούτε ο Γερμανός, το Γάλλος, το Ισπανός ή κανείς άλλος θα φέρουν αντιρρήσεις. Και έτσι όπως του επιτρέπει το Συμβούλιο μπορεί, του επιτρέπει η συνθήκη, το Συμβούλιο μπορεί να επικυρώσει μια υποψηφιότητα παρότι το Κοινοβούλιο έχει εκφέρει αντίθετη γνώμη. Και άρα ναι, μπορούμε να πούμε ότι έχετε ε, σημαντικές δεξιότητες δημοσιονομικό ελεγχτή δεν είσαστε έστω αυτό είναι κάτι που μπορεί να μάθει κανείς εγώ σε αυτό δεν ανησυχώ ιδιαίτερος φαντάζομαι ότι κάποια στιγμή θα γίνεται καλό μέλος του ελεγκτικού συνεδρίου αλλά έχοντας διαβάσει τις προτάσεις κυρία Αγιάλα εξαίρεται στην εκθεσή της δεν θέλω να πω ότι μπορεί να μα λέτε ότι δεν μπορούμε να αλλάξουμε κανόνε. Θα σα διαβεβαιώσω όμω από πλευρά μου ότι εμεί θα του αλλάξουμε του κανόνε και θα ζητήσουμε από του υπουργού μα και κατά πάσα πιθανότητα σε συνεννόηση και συνεργασία με τα εθνικά κοινοβούλια, να αλλάξουν αυτοί οι κανόνες και δεν μας επιβάλλει το Συμβούλιο τους υποψηφίους, γιατί δεν υπάρχει, δεν είναι σωστό αυτό. Εμείς ως Κοινοβούλιο θέλουμε να διορίζουμε τα μέλη του Ελεκτικού Συνεδρίου και να μην έχουμε μόνο γνωμοδότηση. Μας βολεύει λοιπόν αυτό που συνέβη, γιατί μας δίνεται επιχειρήματα. Και τις τροπολογίες μας θα καταθέσουμε, αλλά και η κυρία Γιάλα έχει κάνει καλές προτάσεις, ώστε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ξαναπάρει το πάνω χέρι για τον ε, διορισμό των μελών του ελεκτικού συνεδρίου. Όλα τα ιδιωτικά ε, σώματα δημοσιονομικού ελέγχου, είτε δημόσια είτε ε, ιδιωτικά, πάντοτε δίνουν το δικαίωμα του διορισμού των μελών αυτών στην Γενική Συνέλευση, όχι σε ένα διοικητικό συμβούλιο, δηλαδή σε αντιστοιχεία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και ως εκ τούτου ε, μπορούμε να έχουμε χάρη στη δική σας τάση επιχειρήματα για να διατυπωθούν οι συνθήκες με βέβαια υπογράμμιση των όσων έχουν συμβεί στη δική σας περίπτωση. Και εκ μέρους ομάδας μου, καθώς είμαι και εισηγητή στην ε, περίπτωση που αφορά τη δική σας υποψηφιότητα, ε, όντως συμφωνώ ότι ε, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε, να γυρίσουμε σελίδα. Εκφραστήκατε, είσαστε μέλος πλέον του ελεγκτικού συνεδρίου, αναλάβατε καθήκοντα, αλλά ίσως θα έπρεπε η κυβέρνηση να έχει λάβει υπόψη τις ε, ε, προτάσει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μετά τη δική σα δέσμευση θα έπρεπε να έχει λάβει υπόψη και τη δική σα πρόταση για απόσυρση τη υποψηφιότητά σα και όχι να σα επιβάλλει στο πλαίσιο τη διαδικασία να αναλάβετε καθήκοντα όσο και αν έχει δικαίωμα να το κάνει αυτό ο Πρωθυπουργό. Σε πάση περιπτώσει γυρίζουμε σελίδα λοιπόν και αλλάζουμε τόνο αλλά δεν ε, καταξιώθηκε κανεί ε, με αυτή την στάση. Ευχαριστώ πολύ κύριο Ο Κύριο Στάση έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Λέει ο κύριος Στάς. Κύριε Μάτες, είμαι σίγουρος ότι παρακολουθήσατε τη συζήτηση στην Ολομέλεια που μεταδόθηκε και μάλιστα ζωντανά. Και άκουσα σήμερα τις δηλώσεις σας. Δεν μπορώ να πω ότι αισθάνομαι άνετα μετά από αυτά που άκουσα. Μίλησαν ήδη κάποιοι συνάδελφοι. Δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω μαζί τους. Επίσης, σίγουρα συμφωνώ με τον κύριο Μίλτερ, ο οποίος, ξέρετε, είναι ένας άνθρωπος ε, αμερόληπτος, νυφάλιος, έμπειρος μια που είναι εδώ από το 1994. Και όταν λοιπόν κάποιος του κύριο Μιλντερ λέει τέτοια πράγματα, ε, αυτό σημαίνει ότι μάλλον έχει δίκιο και με τον κύριο Οντι θα συμφωνήσω, ο οποίος μας ανέφερε ότι πήγατε και ήρθατε σε επαφή με τον ε, Πρωθυπουργό σας. Τι γίνεται με την ανεξαρτησία σας και την αμεροληψία σας. Τι να σας μπορείτε τον μεγάλο μουφτή, το, τον Πάπα της Ρώμης ή τον Αυτοκράτορα της Κίνας. Λοιπόν, είδατε, ξέρω εγώ, τον φύλαρχο των Ταλιμπάν, αλλά αυτό τι σχέση έχει με τη δική μας διαδικασία. Τι, τι, να κάνουμε με, με αυτή σας την παρέτηση. Αυτό το οποίο έγινε είναι ότι γυαλ, ράγισε το γυαλί όσον αφορά την εμπιστοσύνη μας προς εμάς. Δεν υπάρχει πλέον η εμπιστοσύνη που προαπαιτείται για αυτά που θέλουμε να κάνουμε και επομένω. Μάλλον με το αριστερό ξεκινάμε την, την συνεργασία μας. Δεν είναι αυτό το οποίο θέλαμε να γίνει. Δεν μπορούν αυτά τα οποία έγιναν να περάσουν έτσι. Ευχαριστώ. Θέλει κάτι άλλο στο λόγο. Όχι, από το βλέπω ο κύριος Γερμπράντη. Αλλά αφού ακούσουμε όλες τις παρεμβάσεις, ήθελα και εγώ ως πρόεδρος να πω κάτι. Εκτός και αν θέλετε να απαντήσετε τώρα στους ακούστηκαν μέχρι στιγμής, κύριε Μάτες. Θα απαντήσετε τώρα ή μετά. Ναι, αν μου επιτρέπετε να απαντήσω τώρα. Η τροποποίηση των κανόνων. Δεν έχω τίποτα κατά μια τέτοια τροποποίηση, αλλά η τροποποίηση θα πρέπει να γίνει βάση των συγκεκριμένων διαδικασιών. Το πρόβλημα που είχα εντοπίσει εγώ είναι ότι ε, όταν θέλετε εκ των, προτέρων να αναλάβουν ορισμένοι άνθρωποι κάποιες θέσεις, δεν είναι δυνατόν να προβλέπετε εκ των υστέρων τροποποίηση των κανόνων. Δεν έχω πάντως τίποτα κατά της τροποποίησης των κανόνων εν γέννη. Πώς κατέληξα στην ε, απόφασή μου να επικυρώσω τελικά το διορισμό μου. Τα εξηγώ όλα αυτά σε μια παράγραφο τη επιστολή μου. Λέω ότι μετά την αρνητική γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ανέλησα την κατάσταση και είδα ότι ιδιαίτερη αιμονή είχε δοθεί στο ζήτημα τη δέσμευση και όχι τόσο στα πραγματικά επαγγελματικά αξιοκρατικά μου προσόντα. Και νομίζω ότι αυτό βάρνε τελικά πολύ περισσότερο. Τα όσα σας είπα δηλαδή στη τελευταία σας ερώτηση βάρναν πολύ περισσότερο από ό,τι στην αξιολόγηση των ικανοτήτων μου. Επιμένατε πάρα πολύ στην ερώτηση αυτή, θέλατε μια απάντηση, σας έδωσα μια απάντηση, έγινε μια συζήτηση και από ό,τι φαίνεται ικανοποίησα πλήρως με την απάντηση αυτή. Πάντως σε κάποια στιγμή όντως είπα τι θα έκανα και όντως για τις επόμενες εβδομάδες μετά την αρνητική γνωμοδότησή σας είχα το στόχο να αποσύρω την υποψηφιότητά μου και γι' αυτό το λόγο πήγα και είδα και τον Πρωθυπουργό μου. Για ποιο λόγο όμω θελήσατε εσείς να είχατε μια τέτοια δήλωση από μένα. Δεν συμφωνούσα τελικά πάρα πολύ με την δική σας τη στάση, με το ότι θέλατε να αποσπάσετε μια τέτοια δήλωση από μένα. Κατά αυτόν τον τρόπο λοιπόν μπορώ να εξηγήσω και την δική μου την τοποθέτηση. Κύριε Πρόεδρε, τι άλλο πρέπει να σας απαντήσω αυτή τη στιγμή. Όχι, μπορείτε να απαντήσετε σε οποιαδήποτε ερώτηση θέλετε. Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι συνάδελφοι που θα να πάρουν το λόγο. Ο κύριος Γκεμπραντή. Κυρία Γιάλα στη συνέχεια. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Αν με ρωτούσατε αν υπάρχει κάτι πιο σημαντικό από τους κανόνες και τις διαδικασίες, τότε θα σας έλεγα ότι εξαρτάται από τις περιστάσεις τελικά. Εξαρτάται από το πεδίο δράσης του καθενός. Αν κάποιος οδηγεί και περάσει με κόκκινο, τότε είναι σαφέστατο το ότι το άτομο αυτό έχει παραβεί τους κανόνες. Και δεν νομίζω ότι είναι συζητήσιμο το θα πρέπει να σας δοθεί πρόστιμο ή όχι. Προφανώς πρέπει να σας δοθεί ένα πρόστιμο, να σε επιβληθεί ένα πρόστιμο. Όσον αφορά την πολιτική, τα πράγματα είναι λίγο πιο ρευστά. Πέρα από τις διαδικασίες, πέρα από τους κανόνες, υπάρχει κάτι πιο σημαντικό. Η εμπιστοσύνη, η αμοιβαία εμπιστοσύνη. Μπορεί κανείς να ακολουθεί πιστά όλους τους κανόνες και όλες τις διαδικασίες, αλλά αν αποσιάσει τελικά η εμπιστοσύνη, τότε το σύστημα δεν λειτουργεί. Νομίζω ότι στην πολιτική αυτό ισχύει. Δεν θα επαναλάβω αυτή τη στιγμή αυτά τα οποία είπαν οι προλαλήσαντες. Ωστόσο, οι σημερινές σας δηλώσεις σε καμία περίπτωση μάλλον αυξάνουν, θα έλεγα, την έλλειψη εμπιστοσύνης και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργούν ή δεν συμβάλλουν στην αποκατασταθη αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη η οποία έχει χαθεί αυτή τη στιγμή. Μία πολύ συγκεκριμένη ερώτηση θα ήθελα να σας υποβάλω. Αν σύμφωνα λοιπόν με τους κανόνες, και όντως αυτό ισχύει, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει δικαίωμα αρνησικηρίας όσον αφορά το διορισμό των νέων μελών του ελεκτικού συνεδρίου. Για ποιο λόγο θεωρείτε εσείς ότι επιμένουμε τόσο πολύ στο να διοργανώνουμε ακροάσεις και άλλες σχετικές διαδικασίες που έχουν να κάνουν με τον διορισμό των νέων μελών του ελεκτικού συνεδρίου. Για ποιο λόγο ασχολούμεθα με τη διαδικασία αυτή, αν δεν είχε κάποια σημασία τελικά. Για να το πω με άλλα λόγια, θεωρείτε ότι αυτό που θα κάνουμε την επόμενη Πέμπτη με τους νέους υποψήφιους είναι τελικά χρήσιμο, εξυπηρετεί κάτι, μήπως θα ήταν καλύτερο να σταματήσει όλη αυτή η παράσταση ε, και ουσιαστικά να αποφασίζει μόνο το Συμβούλιο ή εσείς να παίρνετε μία απόφαση. Θεωρείτε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει πραγματικά κάποιο επικοδομητικό ρόλο. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Ακούσατε όλες αυτές τις παρατηρήσεις από κάποιους ε, πολύ έμπειρους ε, συναδέλφους αυτής της Επιτροπής. Και όταν αναφερόμαστε στο Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι αναφερόμαστε σε ένα θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο ελέγχει τη δημοσιονομική κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ουσιαστικά προχωρεί και στην απαλλαγή. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει ένα ύψιστο επίπεδο λογοδοσίας και εμπιστοσύνης. Και βέβαια και είναι ψηλότατο επίπεδο επαγγελματισμού. Όλα αυτά τα στοιχεία είναι πάρα πολύ σημαντικά για την επιτέλεση των καθηκόντων σας. Και από ό,τι ακούω τώρα από εσά, βλέπω τελικά ότι απαντάτε ιδιαίτερα αποστασιοποιημένα. Λέτε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν επιτελεί κάποιο πολύ σημαντικό ρόλο, δεν έχει τελικά τον τελικό λόγο. Θεωρώ ότι ε, από δημοκρατικής πλευράς δεν αντιδράτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Είπατε επίσης ότι αξιολογήσατε εσείς αρνητικά τη δική μας τη γνωμοδότηση, τις δικές μας παρατηρήσεις. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι η μελλοντική μας συνεργασία θα είναι αρκετά περιορισμένη τελικά και προβληματική. Εμείς δεν θα μας σε θέση να σας υποστηρίξουμε στο έργο σας ως εκπρόσωπο της ε, Κροατίας και βλέπω ότι ήδη το είπατε κι εσείς ότι δεν θα είστε σε θέση, δεν είστε ήδη ανεξάρτητος. Αυτό φαίνεται από την σχέση που έχετε με τον Πρωθυπουργό σας. Δεν ξέρω αν στην επιτέλεση των καθηκόντα σα στα πλαίσια του ελεκτικού συνεδρίου θα συνεχίσετε να προστατεύετε απλώ τα συμφέροντα τη κυβέρνησή σα. Πώ πιστεύετε λοιπόν ότι μπορούμε να έχουμε μια πραγματικά επικοδομητική συνεργασία. Όταν για παράδειγμα εσείς θα υποβάλλετε μια έκθεση, θα μπορούμε εμείς ποτέ να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι η έκθεση αυτή είναι άρτια, ότι είναι άξια εμπιστοσύνης μετά όλες αυτές τις δηλώσεις που κάνατε. Πώς βλέπετε εσείς να διαμορφώνεται η μεταξύ μόν μελλοντική συνεργασία. Γιατί θα πρέπει να γνωρίζετε ότι ο Πρωθυπουργό της ε, Κροατίας δεν θα σας προστατεύει πάντα. Παρακαλώ κύριε Μάτες, για να δούμε. Τίποτα από τα όσα είπα δεν ε, υπενήσεται ότι υποτιμώ το ρόλο του Κοινοβουλίου στη διαδικασία. Δεν εννοώ τίποτα σχετικό. Το προσπαθώ να πω είναι ότι ο ρόλος αυτός υποβιβάζεται αν συνδεθεί με τη συζήτηση περί δέσμευση ενός υποψηφίου να αποσύρει την υποψηφιότητά του. Επηρεάζεται δηλαδή αρνητικά η δυνατότητα σας να επηρεάσετε την τελική απόφαση. Εάν δηλαδή επικεντρωνόσασταν στην αξιολόγηση των ικανοτήτων, των προσόντων των υποψηφίων και δεν περιορίζασταν σε ένα μόνο ναι ή όχι και δίνατε μια έκθεση με δύο-τρεις σελίδες για το λόγο για τον οποίο υποστηρίζεται ή όχι ένας υποψήφιος, κάτι τέτοιο πιστεύω θα ενίσχυε σημαντικά την επίδραση αυτής της αποφασής. Τις προτάσεις κάνουν τα κράτη-μέλη ουσιαστικά. Και όταν ένα κράτο ε, κάνει μια πρόταση θα θέλει περισσότερο από ένα απλό ναι ή όχι. Θα ήθελε μια εξήγηση γιατί και πώς αξιολογείται με βάση τα κριτήρια της συνθήκης ή με την πρακτική που έχει ακολουθεί τα τελευταία χρόνια η παρουσία ενός ψηφίου. Εγώ δεν λέω ότι πρέπει να έχει ρόλο στη διαδικασία το Κοινοβούλιο. και νομίζω ότι επηρεάζεται αρνητικά το, η θέση του κοινοβουλίου από τη στάση αυτή. Για τις εκθέσεις φαντάζομαι ότι θα τις αξιολογείτε με τη βάση των όσων περιλαμβάνουν γραπτός. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να ε, υποβάλω προτάσεις πιστικές. Και βεβαίως και εσείς θα κρίνετε τι θέλετε να διαβάσετε. Θα κάνω ό,τι μπορώ να καταθέτω καλές προτάσεις. Αυτό έχω να πω με τις εκθέσεις μου. Σας ευχαριστώ. Κυρία Αγιάλα Σέντερ και μετά κυρία Γκρέσλε. Κύριε Πρόεδρε, όσοι εισηγήτρια, εάν μου επιτρέπετε, θα προτιμούσα να λάβω το λόγο τελευταία. Κυρία Γκρέσλε, σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να διασκεδάσω λίγο την εντύπωση ότι εδώ το θέμα μας είναι ο κύριος Μάτες. Όχι, το θέμα μας είναι η σχέση μας με το Συμβούλιο. Και παρακολουθούμε ασφαλώς, παρακολουθούμαστε από αρκετό κοινό μέσω των ε, ηλεκτρονικών υπολογιστών. Κύριε Μάτες, τώρα εσείς ε, έχετε ανεβάσει πολύ τον πύχη σε σχέση με προσεχείς υποψηφίους. Θα είναι πολύ πιο δύσκολο και δυσάρεστο να διαπραγματευτούμε με, επόμενου επόμενους μετά από σας υποψηφίους. Αλλά πρέπει να σας πω ότι πάντοτε θα πρέπει αυτό να κάνουμε. Δεν, έχει, δεν θα είναι ποτέ δηλαδή κάτι το εύκολο. Ούτε και ήσασταν μια απλή παρένθεση η δική σας περίπτωση. Πάντοτε έτσι θα συμπεριφερόμαστε. Και πρέπει αυτό να το κάνουμε για να δείξουμε και ότι έχουμε τις απόψεις μας και τις ακολουθούμε. Και πρέπει πάλι να κοιτάξουμε προς το μέλλον, το οποίο δεν φαίνεται τόσο εύκολο. Έχουμε το Συμβούλιο, το οποίο έχει μια νομική θέση γνωστή της πάση, αλλά υπάρχουν και στοιχεία τα οποία ενισχύουν τη θέση του Συμβουλίου, γιατί έχουμε ιστορικά ε, αρκετά κακές σχέσεις με το Συμβούλιο και όχι μόνο για τα οικονομικά στοιχεία, για τα αριθμητικά στοιχεία, αλλά και στην ουσία των σχέσεων μας. Εκ μέρους του ΕΛΚ πάντως εγώ σας, θα σας υπόσχομαι ότι δεν πρόκειται να αφήσουμε σε, σε χλωρό κλαρί το ελεγκτικό συνέδριο πλέον θα παρακολουθούμε τα peer reviews, θα παρακολουθούμε ενδεχόμενο προστασίας κρατών μελών από άλλα κράτη-μέλη, θα παρακολουθούμε πώς γίνονται οι μεταφορές κονδυλίων από τη μια εκθέση στην άλλη και από τη μια στήλη στην άλλη. Δεν πρόκειται να αφήσουμε κανέναν σε χλωρό κλαρί από εδώ και μπρος, σας διαβεβαιούμε. Και φυσικά καλό θα ήταν να συζητήσουμε τα θέματα αυτά ουσιαστικά γιατί το ζήτημα είναι η αποτελεσματικότητα του ελεγκτικού συνεδρίου, τα αποτελέσματα στην λειτουργία του και οι σχέσεις συνεργασίας μεταξύ των θεσμικών οργάνων και του Συμβουλίου βέβαια και του Κοινοβουλίου και οι σχέσεις των μέλων του ελεγκτικού συνεδρίου με την κυβέρνηση, της, ε, με την κυβέρνηση, εν προκειμένου τη δική σας. Θα δούμε λοιπόν πώς θα είναι αυτές οι σχέσεις στο μέλλον. Πάντως, μέχρι τώρα είχαμε καλή ε, διάθεση στην ιστορία αυτή. Για μένα εδώ τελειώνει η καλή διάθεση και καλές προθέσεις. Δεν θα συνεχίσω έτσι και θα συζητούμε τα πράγματα τα οποία είναι πραγματικά σημαντικά, δομικά σημαντικά ε, για την περαιτέρω συνεργασία. Ευχαριστώ πολύ κυρία Γκρέτσλε. Θέλετε να απαντήσετε σε αυτό αμέσως κύριε Μάτης, δεν είστε υποχρεωμένος. Πριν δώσω το λόγο στην συγγήτρια για να δώσω τα δικά της συμπεράσματα, θα ήθελα εγώ και ολοκληρώνοντας τα όσα ακούστηκαν και συνοψίζοντας, αλλά και ως πρόεδρος για να πω δύο λόγια, να πω ποια είναι τα ζητήματα προκύπτουν, κατά τη δική μου έποψη. Καταρχάς έχουμε μια διαδικασία ακρόασης που αποτελεί τμήμα του, της διαδικασίας ορισμού ε, ενός μέλους του ελεγκτικού συνέδριου εκ μέρους του Κοινοβουλίου. Εάν δεν έχει καμία βαρύτητα αυτή η διαδικασία των ακρεάσεων, τίθεται το ερώτημα τι είδους δημοκρατικό έλεγχο μπορούμε να έχουμε και τι σημαίνει δημοκρατικός έλεγχος. Εμείς είμαστε και θεωρούμε ότι είμαστε το άμεσα εκλεγμένο κοινοβουλευτικό σώμα, εκλεγμένο από τον πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είμαστε το κοινοβούλιο, άλλωστε, άλλωστε το εξέφρασαν και αρκετοί συνάδελφοι, το οποίο μπορεί ως άμεσα ερετό σώμα να και οφείλει να διαμορφώσει μία γνώμη για έναν υποψήφιο, μία υποψήφια, τις ικανότητες αλλά και τον χαρακτήρα και την συμπεριφορά της τάσης του δηλαδή έναντι ενός τέτοιου ε, ε, ρόλου, μιας θέσεως και των καθηκόντων που απορρέουν από αυτή. Και ως εκ τούτου αυτή η γνώμη που διαμορφώνουμε μπορεί και οφείλει να ληφθεί η πλήρωση υπόψη μέσα σε κάθε αίσθημα ευθύνη βεβαίω που έχει το Κοινοβούλιο στην απόφαση που θα λάβει. Ο Σάρφος Μιούλντερ μας επισημαίνει επίσης ότι ήταν σημαντική η πλειοψηφία τη Ολομέλεια και όχι μια ασιασδήποτε επιτροπή, τη Ολομέλεια του Κοινοβουλίου, η οποία έχει απορρίψει την υποψηφιότητα του κυρίου Μάτες και αυτό είναι γεγονός. Σήμερα μας ε, καταστήσατε σαφές ότι οι δηλώσεις ενώπιον της Επιτροπής και μέσω αυτής ενώπιον ολόκληρου του Κοινοβουλίου και ουσιαστικά μέσω του Κοινοβουλίου οι δηλώσεις προς όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι δηλώσεις λοιπόν έναντι του ερετού κοινοβουλευτικού οργάνου που εκπροσωπεί όλου του πολίτε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, απεσύρθησαν. Τις δώσατε διαβεβαιώσει, τι οποίε αποσύρατε. Μα είπατε ότι τηρήσατε την υπόσχεσή σα στον βαθμό που προτείνατε την απαραίτητη σα προ την κυβέρνησή σα. και ζητήσατε συγγνώμη για το ότι δεν τηρήσατε την υπόσχεση αυτή προ την Επιτροπή μας. Εάν η Επιτροπή μας τώρα θεωρεί επαρκή τη συγγνώμη αυτή και αν εν γέννη αυτή η δυσάρεστη υπόθεση είναι κάτι που μπορούμε να ξεχάσουμε, δεν θα κλείσει σήμερα, είναι κάτι που δεν θα κλείσει σήμερα. Ίσως χρειαστεί να το συζητήσουν και οι ομάδες και να ληφθεί υπόψη και σε άλλα κέντρα αποφάσεων και σε άλλα σημεία αυτή η υπόθεση. Πάντως θέλω να είμαστε βέβαιοι ότι σας έχουμε καταλάβει καλά. Εξηγήσαμε. Μας εξηγήσετε μάλλον ότι δεδομένη στις δέσμευσεις που είχατε λάβει και τις αποφάσεις που λάβαμε εμείς, ε, την, δηλώσατε την πρόθεσή σας να υποβάλλετε παρέτηση στην κυβέρνησή σας, όμως η κυβέρνηση σας είπε όχι δεν πρέπει να υποβάλλεις παρέτηση και εξωτού ανακαλέσατε αυτήν την δέσμευση και ε, άρα δεν ε, τηρήσατε την υπόσχεση αυτή ενώπιον του δημοκρατικά εκλεγμένου κοινοβουλίου. Τώρα φαντάζεστε τι εικόνα δίνει το να, κάνει, να λαμβάνει κανείς δεσμεύσει ενώπιον ενός κοινοβουλευτικού οργάνου, ενός κοινοβουλίου και να την ανακαλεί μετά ή να μην την τηρεί, να παραβιάσει τη δεσμευσή του. Τι είδου αξιοπιστία δείχνει για τον ε, ε, υποψήφιο αυτόν και δεν θέλω αυτό να σας επισημάνω ότι μας φαίνεται σε μια πολύ δύσκολη θέση και δύσκολη θέση η οποία ξεπερνά την ιανδήποτε συνθήκη γιατί η αξιοπιστία δεν είναι ζήτημα των συνθήκων, είναι ζήτημα της αξιοπιστίας. Εάν δηλαδή ο λόγος ενός μέλους του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο λόγος που δίνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ισχύει ή δεν ισχύει. Εγώ εδώ ως πρόεδρος Επιτροπής δεσμεύομαι σημειώνω ότι θέλετε να ζητήσετε συγγνώμη στην υπόθεση αυτή. Είναι μια δύσκολη κατάσταση και εσάς. Ήρθατε, θεωρούσατε ότι πρέπει να έρθετε να εξηγήσετε τα κίνητρα που σας οδήγησαν στην επιλογή αυτή. Είναι κάτι που πρέπει να ληφθεί υπόψη, αλλά δεν μπορώ ε, να ε, θεωρήσω ότι εκφράζω τους συναδέλφους λέγοντας ότι γίνεται δεκτή αυτή η συγγνώμη. Νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση και πολύ δυσάρεστη για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Διότι είναι πολύ δυσάρεστο να έχει ληφθεί μια απόφαση με τόσο μεγάλη προψηφία εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να μην τηρηθεί η επαγόμενη από αυτήν δέσμευση περί απόσταση της υποψηφιότητας. Εν πάση περιπτώσει σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας, για το τι ήρθατε εδώ σήμερα το απόγευμα. Δεν ξέρω τι είδου συμπεράσματα μπορεί εδώ και τώρα να διατυπώσει η εισηγήτρια ε, σε σχέση με τις επαφές και τις θεσμικές σχέσεις με το ελεγκτικό συνέδριο φαντάζομαι ότι θα πρέπει να συστήσουμε σε άλλο χρονικό σημείο Είναι κάτι το οποίο όμως θα πρέπει να εξετάσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ασφαλώς και στις διακοινοβουλευτικές μας επαφές με συναδέλφους από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Αλλά και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να επιδιώξουμε μια συνένεση, μια συνεννόηση με τους συναδέλφους από τα Εθνικά Κοινοβούλια για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να αντιμετωπίζονται αυτά τα ζητήματα. Αυτά από πλευρά μου. Η κυρία Γιάννα Σέντερ όμως για να καταλήξουμε στο θέμα αυτό. Παρακαλώ. Ε, με συγχωρείτε, θέλετε να πείτε εσείς κάτι. Κύριε Μάτς, πρώτα. Στο τέλος, λέει ο κύριος Μάτσα. Σε εμά τον τελευταίο λόγο έχει πάντα η συγγήτρια. Σας ευχαριστώ που με καλέσατε κύριε Πρόεδρε και επίσης ε, εκτιμώ πάρα πολύ το πνεύμα της συνεργασία που σας διαπνέει, το πώς ε, έγινε όλη αυτή η διαδρομή για κατέληξουμε στη σημερινή συνάντηση, γιατί θεωρώ ότι αυτό είναι καλός γιονός δια το μέλλον. Και εγώ θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου, τόσο ώστε να συνεργαστώ στο ίδιο πνεύμα όπως συνεργαστήκαμε μέχρι σήμερα και στο μέλλον. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και τώρα για τις καταλητικές παρατηρήσεις θα δώσουμε τώρα την σκητάλη στην κυρία Ινές Αγιάλα Σέντερ. Θα ήθελα κύριε Πρόεδρε πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους συναδέλφους όλους για για τις απόψεις τις οποίες εξέφρασαν, κάτι το οποίο αναβαθμίζει την συζήτησή μας. Ε, και κυρίω, όχι μόνο για την παρούσα φάση διαδικασία, αλλά κυρίω και γενικότερα για τη σχέση με το ελληνικό συνέδριο. Οπότε, κύριε Μάτε, θα πρέπει να μην ξεχνούμε ότι το πρόβλημα δεν ήταν πρόβλημα συγκεκριμένη κυβέρνηση, ήταν θεσμικού χαρακτήρα οι σχέση μα με το Συμβούλιο. Ακριβώ όπω το Συμβούλιο ε, προτείνει, κατεβάζει, διαμορφώνει τις υποψηφιότητες. Ενώ εμείς θέλουμε κάτι να πούμε. Δεν θέλουμε να γίνονται έτσι εικονικά αυτές οι, οι ακροάσεις. Θέλουμε να έχουν ειδικό βάρος, να γέρνουν την πλάστιγκα οι απόψεις μας. Οπότε γι' αυτό σας λέω ότι ε, η ερώτηση, η τελευταία, η ακρότελευταία δεν είναι ε, τυπική. Είναι πάρα πολύ σημαντική όσον αφορά την διακυβέρνηση, όσον αφορά εμάς. Εσείς δεν μπορέσατε να κατανοήσετε το πόσο σημαντική ήταν αυτή η ερώτηση για εμάς στο Κοινοβούλιο. Το πρόβλημα δεν είναι η κυβέρνησή σας. Το πρόβλημα είναι κατά κάποιο τρόπο εσείς πώς βιώσατε αυτό το οποίο έγινε συνειδησιακά ας το πούμε. Αυτό που είπατε, η συνείδησή σας και ζητήσατε αυτή την παρέτηση. Οπότε και γι' αυτό το λόγο ε, κατά τη δική μου προσωπικά άποψη τουλάχιστον, όλα αυτά να αμφιβόλο την σχέση εμπιστοσύνη που έχουμε. Και τέλος πάντων ακούσαμε ε, όλα αυτά τα, τα συμβαστικά από τους συναδέλφους, ακούσαμε άλλα ε, σύμφωνα με τα οποία διατύπωσαν κάποιε επιφυλάξει. Εμεί δεν θέλουμε να γίνουν ακόμα πιο ευάλωτε. Να μην, μην γελίσει ακόμα περισσότερο το γέλιο τη με το ελεκτικό συνέδριο. Οπότε τουλάχιστον ξεράγουμε κάποια συμπεράσματα, κάποια μαθήματα από αυτά το οποία έγιναν. Ε, γιατί είδατε τι έγινε. Ε, είδατε η συνείδησή σα που σα ε, οδήγησε. Γιατί αυτή η ερώτηση που δεν καταλάβατε, γιατί υπευλήθη, υπευλήθη, είναι πάρα πολύ σημαντική για αυτό το κοινοβούλιο. Και γι' αυτό και μα ενδιαφέρει πάρα πολύ να ακούσουμε την απάντηση για να μπορέσουμε να αφογκραστούμε τη, τη, τη, τη, στάση, το, πνεύμα, τη, τι, δυνατότητε τελικά. Το που φτάνουν τελικά τα μελτιών του συνεδρίου, κύριε Μάτες. Οπότε, Εμεί. έτσι, επιτυχώς των όσων έγιναν τώρα θα υποβάλουμε την έκθεσή μας, θα συνεχίσουμε τη μάχη που δίνουμε με το Συμβούλιο όσον αφορά τις υποψηφιότητες, ούτως ώστε οι υποψηφιότητε, να είναι αυτές που πρέπει, να είναι πιο δόκιμες για το ελληνικό συνέδριο. Οπότε, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε και, κατακλείδη, θέλω να σα πω ότι το βιογραφικό δεν αρκεί. Χρειάζεται και μια στάση συνεργασίας, κατανόησης, δηλαδή αυτό πάει να πει εμπιστοσύνη από και προς ένα θεσμικό όργανο προς το Κοινοβούλιο, το οποίο πολλές φορές βρίσκεται απέναντι, βρίσκεται να κοντράρει άλλα θεσμικά όργανα. Επομένως αυτό που χρειάζεται είναι να υπάρχει βάθος κατανόηση του τι πάει να πει ε, διακυβέρνηση. Αυτό που να ξέρετε υποψήφι. Δεν αρκεί να ξέρετε απ' έξω τι συνθήκη και τα άρθρα της. Χρειάζεται να ξέρετε τι σημαίνουν, πώς λειτουργούν, γιατί έτσι χτίστηκε η Ευρώπη και το Κοινοβούλιο με αυτές τις μικρές ερωτησούλες, οι οποίες όμως ακριβώς μας οδηγούν σε αυτές τις εγγύσεις, την εγγύση που μας προσφέρει η EMB στο ΣΥΝΙ. κάποια στιγμή θα θέλαμε να φτάσουμε ε, στο σημείο κατά το οποίο να μην επιβάλλονται, να μην προτείνονται από τις κυβερνήσεις υποψηφιότητες για τέτοιες θέσει. Έτσι. Θα έχουμε και καλύτερο ελεγκτικό συνέδριο και καλύτερο έλεγχο του προπολογισμού. Σας εύχομαι πάντως καλή επιτυχία. Και επίσης οι σχέσεις σας με το Κοινοβούλιο και με τα θεσμικά όργανα πάντα γίνονται επ' αυτής της βάσης. Και όχι επ' της βάσης των σχέσεων με την κυβέρνησή σας. Αποδεχόμαστε τη συγγνώμη σας, αλλά παρακαλώ λάβετε όλα αυτά τα οποία είπαμε υπόψη για το μέλλον. Ο Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ κύριε Κερασέντερ. Ευχαριστώ κύριε Μάτες που ήρθατε μέχρι εδώ. Στο σημείο αυτό διακόπτω τη συνεδρίαση. Αύριο συνεχίζουμε στις 9 το πρωί πάλι με δημόσια συνεδρίαση. Ευχαριστώ πολύ.